παρέμβαση της κυρίας Κιέγκε, παρακαλώ. Ο συνάδελφος Μωράης, παρακαλώ. Chairman, um, Κύριε Πρόεδρε, με βάση το 11.2 τον κανόνα που αφορά τη συμπεριφορά των Ευρωβουλευτών που θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμοιβαίο σεβασμό με βάση τις αρχές ε, και τις αξίες ε, των βασικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε από τον κύριο Γιάννου Κόρβιν Μίκε στην προηγούμενη συζήτηση απαράδεκτα σχόλια, απαράδεκτα για το ύφος και το κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, έκανε αντισημητικά σχόλια ο κύριος Κόρβιν Μίκε και φαντάζομαι ότι πολλοί ευρωβουλευτές ε, διαμαρτυρήθηκαν. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθεί δράση, κατάλληλη δράση από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να γίνουν τα σωστά διαβήματα. Και μάλιστα η κυρία Σεσίλ Κέγκε, παρακαθήμενη, υπέβαλε τέτοια σχόλια και θα ήθελε να κάνει και κάποιες συμπληρωματικέ παρατηρήσεις. Frau Κύριε Πρόεδρε, Αναφέρομαι επίση και εγώ στην αναφορά που έκανε ο συνάδελφο αυτό σήμερα το πρωί. Με τι δηλώσει που έκανε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πραγματικά προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του σώματο αυτού. Την αξιοπρέπεια του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, λοιπόν, καθώ επίση και το ίδιο το πνεύμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι οι δηλώσει που έκανε πραγματικά αντιτίθενται στο άρθρο 11, σημείο 2 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δηλώσεις που έκανε δεν προσέβαλαν μόνο άτομα σαν εμένα, που έχουμε διαφορετικό χρώμα δέρματος, αλλά ουσιαστικά προσβάλλουν και όλους αυτούς οι οποίοι εντάσσονται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιτάσσονται οι δηλώσει βασικέ αρχέ τη ισότητα των πολιτών, των ανθρώπων. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να επιβληθούν οι κατάλληλε κυρώσει στον άνθρωπο αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι αναφορέ, τα σχόλια τα οποία γίνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν από εδώ, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ξεκινήσει ένα πραγματικό αγώνα κατά του ρατσισμού. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Κιέγκε. Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έχει ενημερωθεί για αυτό το γεγονός. Επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξης, δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής που αφορούν ε, τη, σε σχέση με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και την καταβολή ε, κονδυλίων και ποσών. Δεν μπορώ να λάβω διαδικαστικό για αυτό το θέμα πλέον. Λυπούμε. Μια ερώτηση λέτε. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Παρεμβάσεις επιθεμάτων επί των οποίων πρέπει να πω συμμερίζομαι επί του περιεχομένου αλλά να μην αφήσουμε τα πράγματα να πείτε ότι ενημερωθήκατε για αυτό το συμβάν αλλά να επισημάνετε ότι θα αναλυφθεί κάποια δράση κάποιο διάβημα για αυτά τα γεγονότα. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε πώς δρούμε εδώ στο σώμα. Ο πρόεδρος ενημερώθηκε για αυτό το γεγονός. Είναι δική του αρμοδιότητα να συναγάγει συμπεράσματα που ενδεχόμενα θα οδηγήσουν και στην επιβολή κυρώσεων. Γι' αυτό το είπα αυτό το οποίο